όλα να δώσω το λόγο στους ε, συντάκτες. Ε, ξεκινάμε με τον ε, κύριο Αλμπρέχτη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε σήμερα για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Νομίζω λοιπόν ότι έχει φτάσει πλέον η χρονική στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, πέρα από τις ε, πολιτικές ομάδες, εμείς καταθέσαμε μία επερώτηση αναφέροντας ε, ότι η μεταρρύθμιση του εντάλματος αυτού και η εφαρμογή του επίσης αμφισβητούνται. Παρακαλούμε λοιπόν την Κομισιόν και το, Συμβούλιο να καταθέσουν προτάσεις. Το Ευρωπαϊκό πρόβλημα σύλληψης ε, ήταν κάτι που υποτίθεται θα γινόταν στο πλαίσιο της αναγνώρισης των διαφορετικών συστημάτων δικαίου. Όταν λοιπόν εγκρίθηκε αυτό το ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο μιας απόφασης πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κατέστησε σαφές ότι τα κριτήρια είναι αρκετά υψηλά, δηλαδή το ένταλμα θα ισχύει μόνο για αυστηρές ποινές, ε, για εγκλήματα, κακουργήματα και πάνω και ότι θα πρέπει να ε, εναρμονιστούν οι διαδικασίες. Ε, δυστυχώς η εναρμόνιση αυτή δεν έλαβε χώρα τουλάχιστον όχι κατά 100%. Υπάρχουν πάρα πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις και σε αυτές βλέπουμε ότι αυτό που σας είπα ισχύει, δεν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει προσαρμογή και στην πρακτική και στις νομοθεσίες. Ελπίζω στην εναρμόνιση των διαδικασιών τώρα μετά από 10 χρόνια ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με τη βοήθεια της κυρίας Ρέντινγκ. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να κάνουμε πάρα πολλά βήματα και στις ε, συνθήκες κράτησης αλλά και στο θέμα ε, των εγγυήσεων προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι μόνο να προχωρήσουμε στην περαιτέρω αναγνώριση των αστυνομικών αρχών και τη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και σε θέματα ποινική δικονομίας. Θέλω να πιστεύω ότι το ένταλμα σύλληψη ε, πρέπει να προσαρμοστεί γιατί δεν είναι πλέον συμβατό με τα κριτήρια που είχαμε εμείς ε, απαιτήσει, δηλαδή να ε, κρίνεται το θέμα της αναλογικότητας τουλάχιστον σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Μπουζουτήλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήταν ένα ευρωπαϊκό όργανο αυτό που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα στον τομέα της δικαιοσύνη. Αυτό ήταν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα το οποίο κατήργησε τα σύνορα. Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, λέγοντας ότι αν κάποιος κάνει ένα αδίκημα σε μια χώρα, δεν μπορεί να ξεφύγει σε άλλη χώρα. Και δεν μπορεί να ξεφύγει από το αδίκημά του και θα διωχθεί. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Εντάλμα Σύλληψης αποτελεί ένα καλό μέσον που έχει θετικά αποτελέσματα. Πράγματι έχει και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία είναι απολύτως εμφανή όταν χρησιμοποιείται για δικήματα τα οποία είναι πολύ ασήμαντα ώστε να δικαιολογήσουν τη χρήση του. Δεν περιμένω ότι το ένταλμα θα εκδοθεί αν συλληφθεί κάποιος να κλέβει λάστιχα ενός αυτοκινήτου σε κάποια χώρα όπως έχει συμβεί. Γιατί στην περίπτωση αυτή θα είναι δυσανάλογη η χρήση του και θα αφαιρούσε, θα περιόριζε την εμπιστοσύνη του κόσμου σε ένα σημαντικό και καλό μέσον. Ως εκ τούτου πρέπει να εντοπίσουμε αυτά τα μειονεκτήματα κατά την χρήση και την εφαρμογή του εντάλματος, χωρίς όμως να το καταστρέψουμε και να το καταργήσουμε. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν πρέπει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς έχει εφαρμοστεί τα τελευταία αυτά χρόνια το ένταλμα. Πράγματι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε αν θα πρέπει να αλλάξει για να χρησιμοποιηθεί ως, όπως δει. Λάτφορτ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε υποστήριζε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Γιατί, γιατί είναι σημαντικό στην στον αγώνα μας εναντίον του διασυνοριακού εγκλήματος. Όμως, η ομάδα μας ταυτόχρονα πάντοτε υπογράμμιζε ότι το σύστημα του Ευρωπαϊκού, Συντάγμα, ε, Ευρωπαϊκού Εντάλματος θα ήταν ε, ανεπαρκές αν δεν συνοδευόταν από τα κατάλληλα δικονομικά δικαιώματα ε, στην Ευρωπαϊκή, κοινά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τα δικαιώματα υπεράσπιση αλλάζουν μετά από πρόταση κομισιών και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ρέντινγκ για τον οδικό χάρτη που έχει παρουσιάσει. Το θέμα είναι το εξή. Θα είναι αρκετή αυτή η δράση για να αντισταθμίσει τι αδυναμίε του συστήματο Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Εγώ πιστεύω πω όχι. Γιατί θα πρέπει να δούμε το πώ λειτουργεί το, το ένταλμα. Αναγνωρίζουμε τι επιτυχίε ανάμεσα στο 2005 και 2009 το ένταλμα εξασφάλισε την έκδοση 12.000 κακοποιών, λάθρεπων ναρκωτικών, βιαστών κλπ. Και δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε και στην ε, εξυχνίαση ε, ε, του, του εγκλήματος του, της τρομοκρατικής ενέργειας στο μετρό του, Λονδίνου το 2005 πολλοί Βρετανοί θα, χαιρώνουν, θα πρέπει να χαίρονται ε, παρόλο ότι πολλοί ευρωσκεπτικιστές επικρίνουν το ένταλμα. Το Ενωμένο Βασίλειο βέβαια είναι αλήθεια πως έχει, το, είναι δεύτερη στη λίστα των ε, ετοιμάτων που, δεύτερη στη λίστα των ετοιμάτων που δέχεται για τη χρήση του ε, και έχουν βέβαια γίνει και καταγγελίες για λαθασμένη χρήση του. Για παράδειγμα, χρήση του εντάλματος για ελάσσονο σημασίας αδικήματα, ε, μεγάλες περίοδοι κράτησης πρώτης δίκης και ψηλές επιδικαστέντε αποζημιώσεις, αποζημιώσεις για την προσωρινή απελευθέρωση ε, για ξελουδαπούς πολίτες. Η Κομισιόν δεν φαίνεται ότι είναι υπέρ της αναδιατύπωσης του, αντιστοιχη της αντίστοιχης Εμείς πιστεύουμε πως ναι, πως χρειάζεται. Χρειάζεται μεγαλύτερη, περισσότερη έλεγχη αναλογικότητας ε, δεν θα πρέπει να καλύπτονται τα ελάσσον σημασία αδικήματα. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνεται και ένας ρητός έλεγχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εκτελών κράτος. Ε, ρητός εννοώ, όχι έμεσος. Τρίτον, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ε, εκεί που δεν είναι λογικό να εκτελεστεί ένα ένταλμα, σε αυτές τις περιπτώσεις να μην γίνεται έκδοση. και όταν απορριφθεί μια φορά το αίτημα να ε, θεωρείται ότι έχει απορριφθεί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης παρόλο ότι ε, στη βάση του είναι πετυχημένο. Αυτοί που το επικρίνουν ε, θα ήταν ικανοποιημένοι με, με την κατάσταση σύμφωνα με την οποία διάφοροι εγκληματίε θα γυρνούσαν ελεύθερη αριστερά-δεξιά σε διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή οι διαδικασίε έκδοση κατά τα άλλα ήταν πολύ αργέ. Σίπελ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στη συζήτηση που μόλις ολοκληρώθηκε για το Ουγγρικό Σύνταγμα επικρίναμε το ότι η συζήτηση ήταν πολιτικής φύσεως και αυτό με εκπλήσει διότι οι πολιτικές συζητήσεις ε, είναι σαφώς καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα ξεκινήσω με την πολιτική διάσταση του θέματος που συζητάμε. Ε, το οργανωμένο έγκλημα ποτέ δεν σταμάτησε στα σύνορα ούτε την εμπόδιση την εγκληματικότητα αυτή οποιοδήποτε μορφής έλεγχος ε, δεν πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε προβλήματα στη συμβίωση των λαών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο η συνεργασία. Χρειαζόμαστε τη διασυνοριακή συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη αποδείχθηκε επανειλημμένα ένα ιδιαίτερα επιτυχέ εργαλείο. Βέβαια το εργαλείο αυτό δυσφημείται όταν α πούμε εκδίδεται Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη απλά και μόνο επειδή κάποιο έκλεψε ένα ποδήλατο. Ε, Δυστυχώ είμαστε αναγκασμένοι όμω να πούμε ότι να γίνεται κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει, υπάρξει τέτοιε περιπτώσει. Ε, όταν όμως ε, δεν εκδίδεται ένταλμα σύλληψης παρότι υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν σε ότι θα έπρεπε να εκδοθεί αυτό αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση όπου πολίτες ε, διαμαρτύρονται και αυτό σίγουρα δεν συμβάλλει στην αξιοπιστία του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος. Πού οφείλονται όλα αυτά. Μήπως το κείμενο της οδηγίας αφήνει πολύ μεγάλο περιθώριο λιγμών. Μήπως τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά το ένταλμα. Μήπως δεν υπάρχουν οι επαρκείς πληροφορίες. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιωθούν και η Κομισιόν πρέπει να λάβει μέτρα για να παρεμποδίζει τέτοιου είδους αρνητικές ε, καταστάσεις γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε ένα τέτοιο εργαλείο να μην ζημιώνεται και να μην μειώνεται η εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτό. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με το χάρτη πορείας ε, για, τα, ε, για θέματα ποινική δικονομίας. Ε, οι διαδικασίες ποινική δικονομίας θα πρέπει να είναι οι ίδιες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται λοιπόν να αντιμετωπίσει όλες τις αντιδράσεις που προκύπτουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμφίβολα μπορεί και να υπολογίζει στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Σίπελτ, δέχεστε μπλε κάρτα. Πολύ ωραία. Κυρία Σίπελ, περιγράψατε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως μωρό. Μήπως Δε, μήπως θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα τέρας του Frankenstein. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω στην ερώτηση. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Αυτό είναι επίθεση, πολεμική επίθεση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη είναι το κατάλληλο μέσο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το έγκλημα στον ευρωπαϊκό χώρο. Το έγκλημα δεν είναι εθνικό, είναι διεθνέ, είναι διασυνοριακό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε. Ε, τα αρχικά προβλήματα που υπήρξαν με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί και αποδείχθηκε ότι το ένταλμα αυτό είναι εκ των όνου κάνευ. Μπάτεν, τρία λεπτά. Από το 2004 είχα προειδοποίησει ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όργανο καταπίεσης πολιτικά διαφωνούντων. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περίπτωση του Julian Assange. Υπάρχουν πολλές παρατηρηπίες στην περίπτωση στην περίπτωσή του δεν έχει ακόμα κατηγορηθεί για κανένα συγκεκριμένο αδίκημα. Πλήρη, προηγούμενη έρευνα εναντίον του για αυτό που οι Σουηδοί ε, αναφέρουν ως ε, βιασ, ε, ε σε, δεύτερο σε ε, μικρό βαθμό έχει οδηγήσει σε μια ολόκληρη διαδικασία που ε, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Υπάρχει η δυνατότητα να απαλλαγεί ο κύριος Ασάνς. Ανεξάρτητα από αυτό λένε ότι οι κατηγορίες κατά του κυρίου Ασάνς δεν θα μπορούσαν να σταθούν στο, Ευρωπαϊκό, στο Βρετανικό Δικαστήριο. Ε, στη Σουηδία ένας δικηγόρος λέει ότι δεν μπορούν οι ίδιες οι γυναίκες να πούν αν οι πράξεις αυτές συνιστούν βιασμό γιατί δεν είναι δικηγόροι. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει καθορισμός ή εξήγηση του τι, ποιο είναι το αδίκημά του. Ο κύριος Ασάνς παρέμεινε στην ε, Σουηδία για πέντε εβδομάδες για να απαντήσει σε αυτές τις ε, ε, κατηγορίες, αλλά ποτέ δεν το ετέθη ερώτημα. Είχε πάει στην Σουηδία τουλάχιστον ένα, λιγότερο από ένα μήνα αφού είχε η Wikileaks διαρρεύσει τα έγγραφα για το Αφγανιστάν. Έχει ζητηθεί να δολοφονηθεί ίσως ή να απαχθεί ο κύριος Ασάνζ γιατί ε, Wikileaks περιγράφεται ως τρομοκρατική οργάνωση. Όλα αυτά συνάδουν με μια πολύ βολική έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος εναντίον τους. Η Σουηδία έχει πολύ καλή στενή σχέση με τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή στοιχείων κλπ. Και αυτό αμφισβητεί την λεγόμενη ουδετερότητα της Σουηδίας. Γιατί λοιπόν να θέλουν οι, οι ΗΠΑ να εκδοθεί στη Σουηδία ο κύριος Ασάνζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να στηρίξουν την υπόθεση εναντίον του και δεν ξέρουν αν μπορούν να τον κατηγορήσουν για οτιδήποτε. Χωρί κατηγορία δεν μπορούν να τον δώσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει όμω κάπου να τον έχουν φυλακίσει καθώ τα προετοιμάζουν όλα αυτά και να τον εμποδίσουν να τον επιστρέψει στην Αυστραλία. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη αποτελεί το τέλειο μέσον. Όπω σα έχω πει επανειλημμένω εδώ, σύμφωνα με αυτό το ε, ε, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, δικαστική παράδοση όπως θα έπρεπε να ονομάζεται είναι πλέον μια γραφειοκρατική διαδικασία. Δεν υπάρχουν πραγματικά πραγματικές διασφαλίσεις. Κατόπιν όλων αυτών θέλω να ρωτήσω το, το Συμβούλιο και την Κομισιόν όχι αν γίνεται κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για πολιτικούς σκοπούς αλλά αν μπορεί να γίνει κατάχρηση. Αν είναι έντιμη θα πρέπει να παραδεχτούν ότι μπορεί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα σας παρακαλώ. Κατά την άποψή μου τα στοιχεία δείχνουν ότι σαφώς αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Τζούλιαν Ασάνζ. Πολύ ωραία, για δύο λεπτά. Το κείμενο της προφορικής ερώτησης ίσως μοιάζει λίγο θεωρητικό ή πεζό, αλλά μιλάει στην πραγματικότητα για τη μοίρα των ανθρώπων, των πολιτών μας. τις κάτω χώρες η κοινή γνώμη σχολιάζει πολύ ε, την περίπτωση ενός ε, Ολλανδού επιχειρηματία που το 1997 κατηγορήθηκε ότι παραβίασε το προλογικό φορολογικό δίκαιο και κρατήθηκε για, τότε για δύο μήνες. Πλήρωσε μια εγγύηση και απελευθερώθηκε. Από τότε δεν ξανά τίποτε. Πέρσι οι Πολωνοί ζήτησαν την έκδοσή του χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Μια μισή εβδομάδα πριν μεταφέρθηκε στην Πολωνία. Αυτός ο κύριος, ο κύριος Φαντίσελντον, μάλιστα, τοποθετήθηκε σε μια βρωμερή φυλακή ε, στις ίδιες κακές συνθήκες που είχε κρατηθεί το 1997 αντίθετα με όλους τους κανόνες και κατά παράβαση πολλών ε, ε δικαιωμάτων του. Μπορεί να ξαναεκδοθεί ε, ένταλμα σύλληψή του, μάλλον εκδόθηκε ξανά ένταλμα σύλληψή του, ξαναπλήρωσε εγγύηση και απελευθερώθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό το σύστημα, οδηγήσει σε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό μα ανισχύει πολύ στην Ολλανδία. Εμεί βασίζουμε τι ελπίδε μα στην Επίτροπο. Κυρία Επίτροπε, θα μπορούσατε να μα δώσετε μερικέ εξηγήσει για την, το πώ εφαρμόζεται η αρχή τη αναλογικότητα. Θα μπορέσετε να μας εγγυηθείτε ότι ε, δίδεται το δικαίωμα της ε, ε υπεράσπισης ε, αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους έχει εκδοθεί ένταλμα. Τι γίνεται με τις χώρες στις οποίες οι συνθήκες κράτησης είναι απάνθρωπες. Δεν θα έπρεπε εκεί να είναι δυνατόν για αυτές τις χώρες να αρνηθεί ε, εκτελούσα χώρα την εκτέλεση του εντάλματος. Πολύ ωραία. Κύρκοπ, δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις ε, θετικές επιπτώσεις που είχε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα στο διασυνοριακό έγκλημα. Μέχρι τώρα συνέβαλε στο να εκδοθούν περίπου 12.000 ε, έμποροι ναρκωτικών, ε, αυτοί που ασχολούνται με την παιδική πορνεία. Βεβαίως χρειάστηκαν μακρόπνοες διαδικασίες υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ελευθερία και αυτό οδηγεί στην επέκταση του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, ποτέ δεν θέλαμε να αντιμετωπίζονται ίσονος σημασίας ε, παραβιάσει όπως το να κλέψει κανεί μια σοκολάτα. Προφανώ όχι. Αυτό όμω που βλέπουμε σήμερα είναι ότι όλε οι πολιτικέ ομάδε και όλε οι εθνικότητε που βρίσκονται εδώ λένε ότι τώρα πλέον έχει φτάσει η στιγμή να αναθεωρήσουμε, να επανεκτιμήσουμε και αν χρειαστεί να τροποποιήσουμε το ένταλμα αυτό. Αναλογικότητα, προστασία και αποζημίωση είναι το κλειδί στη μεταρρύθμιση. Ε, ασχολούμενοι ε, με τον, ε, με τις έρευνες, όσοι ασχολούνται με τις έρευνες καταλήγουν στο ότι δεν πρέπει να γίνουν και πάλι τέτοια λάθη. Οφείλουμε τη νέα νομοθετική πράξη να τη σχεδιάσουμε μην ξεχνώντας τις ελλείψεις του Ευρωπαϊκού εντάλματο Σύλληψης. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ε, συνθήκων ε, κράτησης απαράδεκτων, ε, που δεν δόθηκε. Αυτό που φοβόμαστε είναι ότι θα προχωρήσουμε με το ένταλμα σύλληψης ε, ενώ η βάση αυτή τη στιγμή δεν είναι σταθερή. Πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη και το ένταλμα αυτό να προβλέπεται μόνο για σοβαρές περιπτώσεις ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα ε, διασφαλίζονται και υψηλές προδιαγραφές κατά την χρήση του εντάλματος. Κύριε Κύρκοπ, δέχεστε μία μπλε κάρτα. Θα ήθελα να πω τον κύριο Κιόρκοπ το εξή. Συμφωνεί ότι πρέπει να αναφερθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Σύλληψη. Ε, Πάντω ε, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή σε ευρωπαϊκές έρευνες, ευρωπαϊκό σύστημα ερευνών. Ίσως αυτό να είναι πολύ προχωρημένο. Ή, ή, όμως μήπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μερικοί είναι υπέρ ε, αυτού του συστήματος και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποσυρθούμε. Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία. Μήπως ε, λοιπόν στην περίπτωση αυτή έχουμε πάλι ένα τρίκα των ε, συντηρητικών ε, της Μεγάλης Βρετανίας όπου εδώ ε, τάσσονται κατά ενός πράγματος ενώ στην πατρίδα τους έχουν διαφορετική στάση. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη θέση της Βρετανικής κυβέρνησης τόσο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όσο και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ερευνών εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το διασυνοριακό έγκλημα. Εμείς ήμασταν ήταν θύματα πολλών εγκλημάτων, κυρίως της τρομοκρατίας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και είμαι σίγουρος, ε, συμφωνείτε μαζί μου, ότι πρέπει με αποφασιστικότητα να εξαλείψουμε την τρομοκρατία. Η βία συνοριακή συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουμε. Βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ερευνών πρέπει να εφαρμόζεται πολύ προσεκτικά. Αλλά και μόνο η έννοια, ε, όπως αναφέρεται, ε, δεν φτάνει. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει αλλάξουν οι λεπτομέρειες του συστήματος αυτού, ε, το σύστημα να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Το γεγονός όμως ότι προσχωρήσαμε σε αυτό το σύστημα είναι κάτι το σωστό. Εμείς ε, θέλουμε να ε, βοηθήσουμε έτσι ώστε να, γίνονται, να, να γίνουν σεβαστές οι απόψεις μας. Grazie. La parola ora al ministro Ghiori, prego. Ο λόγος στην Υπουργό Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε, αγαπητά μέλη. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη είναι ένα από τα πιο επιτυχή εργαλεία αμοιβέ αναγνώριση που έχουν υιοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση. Το Συμβούλιο αφιέρωσε πολλή ενέργεια σε αυτό το ζήτημα και μέσω ε, αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής μεταξύ ομοτήμων. Peer evaluation δηλαδή, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια τριών ετών στα κράτη-μέλη. Το απλεονεκτήματα του εντάλματος ε, είναι πολύ περισσότερα από ότι οποιαδήποτε αδυναμία του. Χάρη, στα, στο ένταλμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να μειώσει τους χρόνους παράδοσης πάρα πολύ. Από ένα ως δύο χρόνια πολλές φορές σε ένα ως δύο μήνες. Το προηγούμενο σύστημα έκδοσης ε, ήταν πολύ γραφειοκρατικό, δυσκίνητο και σίγουρα δεν προσαρμοζόταν στον καινούριο κόσμο των ανοιχτών συνόρων και στα, ε, καινούριου τρόπους λειτουργίας του διασυνοριακού εγκλήματος. Στο θέμα της αναλογικότητας, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ελάσσων σημασίας ε, που εκδόθηκε χωρίς λόγο το ένταλμα, αλλά οι αρχές κάθε κράτους μέλους αποφασίζουν για ποιου είδου αδικήματα ξεκινούν τη διαδικασία του εντάλματο. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αντίθετα με την έκδοση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ε, είναι ένα καθαρά δικαστικό ε, ε, σύστημα. Βασίζεται δηλαδή η έκδοσή του σε μια απόφαση δικαστή, δικαστικού λειτουργού και η ο απόφαση αυτή και τα κριτήρια της λαμβάνονται σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Δικαστικής Αρχής. Αν υπάρχει θέμα αναλογικότητας, αυτό δεν προκύπτει από το ίδιο το εργαλείο, από, το, από την απόφαση πλαίσιο δηλαδή για το ένταλμα. Αυτό αποτε, αυτή η έλλειψη αναλογικότητας ενδεχομένως βασίζεται, ε, ε, οφείλεται στον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν το σύστημα σε εθνικό επίπεδο οι δικαστές. Το ε, ένταλμα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται όταν δεν είναι ε, απαραίτητο. Το Συμβούλιο επίσης έχει καλέσει τους ε, χρήστες να ζητούν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις έναντι της έκδοσης εντάλματος, δεδομένης ε, και της ε, ανάγκης να είμαστε πιο, ε, όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται και να χρησιμοποιούμε τα λιγότερο ισχυρά δυνατόν όπλα που διαθέτουμε στο πλωστάσιό μας. Δεν ε, είναι πολύ για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα πληροφορών της Σέγγεν, να εκδίδονται κλητεύσεις για κατάθεση ή να χρησιμοποιείται η ε, απόφαση πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση ε, οικονομικών κυρώσεων και ποινών. Αυτές πάντως τι αποφάσεις σε κάθε περίπτωση θα τι λαμβάνουν οι εκδίδουσες αρχές. το ευρωπαϊκό ένταλμα εκδίδεται κατόπιν ε, τελεσίδικης απόφασης στο κράτος μέλος έκδοσης. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το υλικό που έχει στην άποψή του και τα τεκμήρια που έχει στην άποψή του ο δικαστή. Και δεν θα πρέπει να αγνοούμε και τα θύματα. Στι περισσότερε περιπτώσει τα θύματα των αδικημάτων βρίσκονται στο κράτο μέλο έκδοση και όχι στο κράτο μέλο εκτέλεση. Συνεπώ, ε, καθυστερώντα την δίκη ε, και την εκδίκαση, τα, πλήττονται και τα ίδια τα δικαιώματα των θυμάτων. Η δικαιοσύνη που αργεί είναι ε, αρνησιδικία, ισοδρομή με αρνησιδικία. Ε, και για τα θύματα. Είναι επίση προ όφελο των θυμάτων να επιταχυνθούν οι δίκε έτσι ώστε να τύχουν προστασία στα δικαιώματά τους. Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει ένα οδικό χάρτη που πρότεινε η Ουγγρική Προεδρία για να ενισχυθούν τα δικαιώματα των θυμάτων. Η λύση στο θέμα της αρχής της αναλογικότητας λοιπόν δεν μπορεί να είναι η τροποποίηση των θεμελίων του συστήματος που λειτουργεί καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει βελτιώσει τα προελιότερα συστήματα έκδοσης. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα στην υπεράσπιση, θα ήθελα καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι αντίθετα με την έκδοση, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, επαναλαμβάνω, είναι ένα πλήρω δικαστικό σύστημα, κάτι που από μόνο το αποτελεί σημαντική εγγύηση. Το ένταλμα βασίζεται πάντοτε σε δικαστική απόφαση του στο κράτος ε, έκδοσης και εκτελείται μόνο αν έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση ο κατηγορούμενος έχει εξασφαλισμένα τα δικαιώματα υπεράσπισής του στο κράτος το οποίο θα γίνει δίκη. Αυτό συμμορφώνεται πλήρως με την νομολογία του ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ε, το άτομο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα δεν ε, έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματά του στο εκτελών κρατός μέλος. η απόφαση 2010 του ε, η οδηγία 64 του 2010 προβλέπει ε, δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνίας ε, καθ' όλες τις διαδικασίες προκύπτουν από την εκτέλεση ενός τέτοιου εντάλματος. Επίσης η Κομισιόν έχει προτείνει πρόσφατα οδηγία για τα δικαιώματα στην πληροφόρηση σε ποινικέ διαδικασίες με γραπτή πληροφόρηση που περιλαμβάνει και τις διαδικασίες του εντάλματος χαιρόμαστε για αυτή την πρόταση. Ε, οποιασδήποτε... Ε, βέβαια, ε, προκύπτουν κατηγορίες ότι όταν απορριφθεί ένα τέτοιο ένταλμα δεν διαγράφεται το αίτημα από το, σύστημα πληροφόρησης Schengen. σύστημα πληροφόρησης Schengen, στο σύστημα πληροφόρησης Schengen τη διαγραφή μπορούν να κάνουν οι αρχές οι οποίες εισήγαγαν το, το συγκεκριμένο στοιχείο. Ε, αν ε, απορριφθεί τελεσίδικα το ε, ε, ένταλμα, το άτομο αυτό δεν μπορεί να συλληφθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Όμως, ε, η απόρριψη δεν ακυρώνει το ένταλμα, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, για παράδειγμα, στο στο κράτος μέλος που το έχει εκδώσει και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Αυτό δεν έχει σχέση με το σύστημα του ευρωπαϊκού ε, Αυτό ίσχυε και στο σύστημα εκδόσεων, έκδοση. Τέλος, ό,τι αφορά τις ε, συνθήκες κράτηση. Ασφαλώ και σε ορισμένε περιπτώσει θα πρέπει να βελτιωθούν. Όμω αυτό δεν έχει άμεση σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών τον, του, εκδίδον, του, του κράτους μέλους να διατηρεί τις φυλακές του και τα κρατήρια του σε, στο σωστό επίπεδο και σωστή ποιότητα ανεξαρτήτως αν το άτομο αυτό που θα κρατηθεί έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί με βάση το ένταλμα ή όχι. Το λόγο έχει η Επίτροπος η κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ. Ε, θα ξέρετε ίσως πως η Κομισιόν υιοθέτησε μια έκθεση για την εφαρμογή του εντάλματος ε, στις 11 ε, Απριλίου φέτος η οποία εστιάζει στις θεμελιώδεις πτυχές της λειτουργίας του εντάλματος σύλληψης και τονίζει για πρώτη φορά από όταν κατέστη επιχειρησιακό τον Ιανουάριο του Τεσσερά όχι μόνο τις επιτυχίες του αλλά και τις ελλείψεις του. Πολλά έχουν ήδη υποθεί για τις επιτυχίες. Να αναφέρω μόνο πως μεταξύ 2005 και 2009 περίπου σχεδόν 55.000 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης ε, εκδόθηκαν, γύρω στα 12.000 εκτελέστηκαν και περίπου 60% των ατόμων αυτών συμφώνησαν στην έκδοσή τους. Κατά μέσο όρο για 17 ημέρες χρόνο παράδοσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ήταν 48 ημέρες ο χρόνος έκδοσης. Και προ Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης είχαμε ε, μέσο όρο ένα έτος για έκδοση ατόμου και οπωσδήποτε ενισχύει και η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων. Γι' αυτό νομίζω πως όλοι συμφωνούν εδώ πέρα πως το ένταλμα σύλληψης είναι σημαντικό μέσο σύλληψης εγκληματιών και μέσο για να γίνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα ποινική δικαιοσύνης και χρησιμεύσε σύλληψη των παιδόφιλων και τρομοκρατών. Όμως και αυτό είναι πρόσφατη εξέλιξη, βλέπουμε από το 2007 πως ο αριθμός των ενταλμάτων που εκδίδονται έχει αυξηθεί δραματικά. Σε πολλές, σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν είναι αναλογικός για να εκδοθούν ύποπτοι μικρό πτεσμάτων που έχουν κλέψει ένα ποδήλατο ας πούμε ή ένα γουρουνόπουλο. Αυτό δεν είναι αναγκαίο και μπορεί να βλάψει και την νομοποίηση αυτού του σημαντικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η Κομισιόν ζητά δράση. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν καλεί τα κρατη να εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας όταν εκδίδουν τέτοιο ένταλμα να γεμίσουν τα κενά επίσης ε, εκείνα τα οποία υπάρχουν όταν δεν συμμορφώνουν την νομοθεσία τους με την οδηγία πλαίσιο ε, του εντάλματος. Επίσης, εισαγγελείς και οι λοιπές αρχές δεν θα πρέπει να εκδίδουν εντάλματα για πτέσματα. Και άρα σε ένα εγχειρίδιο το οποίο θα εκδώσουμε θα αναφέρουμε ποιες θα είναι οι γραμμές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται. Επίσης, πριν το τέλος του έτους θα καταθέσουμε προτάσεις για να ενταθεί η εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών, των δικαστικών αρχών για το ένταλμα σύλληψης για να υπάρχει ενιαία εφαρμογή και αποτελεσματικότητα και να γνωρίζουν τις ε, νέες ευρωπαϊκές ρήτες ασφαλείας για τα δικονομικά δικαιώματα. Τον ε, λέμε τη ευκαιρία των οικονομικών δικαιωμάτων. Τονίζουμε επίσης ε, στην έκθεση την σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει ξεκινήσει να εξετάζει τα δικονομικά δικαιώματα των συλληφθέντων. Π.χ. ελάχιστοι κανόνες, δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση, κατά το οποίο είχε ήδη οθετηθεί το 2010, δικαίωμα στην ενημέρωση περί δικαιωμάτων και θα καταλήξουμε σε συμφωνία πάρα πολύ σύντομα βεβαίω. Επίσης, σήμερα υιοθετήσαμε ως Κομισιόν μία πρόταση για τα δικονομικά δικαιώματα για να διασφαλιστεί πρόσβαση σε δικηγόρο και το δικαίωμα ειδοποίησης τρίτου ατόμου όταν κάποιος ε, στερεί την ελευθερία του. Θα συμπεριληφθεί επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο και στα δύο κράτη-μέλη σε περίπτωση ευρωπαϊκού ενταλματοσύλληψης. Οπότε όλα αυτά τα οικονομικά δικαιώματα ισχύουν για το ένταλμα σύλληψης. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να μην συλλέγονται πληροφορίες κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπόπτων. Θα ήθελα επίσης, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο ετέθη από τους συντάκτες της έκθεσης. Η Κομισιόν δεν γνωρίζει ε, στοιχεία για την ε, αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Σουηδία για έκδοση του κυρίου Ασάνζ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων είναι χρήση ε, η οποία δεν είναι σωστή. Πρόκειται, όπως σας είπα, για μια τελείως δικαστική διαδικασία στην οποία οι κυβερνήσεις δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης. Στη δε συγκεκριμένη περίπτωση που ε, αναφέρει το Κοινοβούλιο την υπόθεση έχουν αναλάβει οι δικαστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας χωρίς την παρέμβαση κυβερνήσεων. Τα, το άλλο ερώτημα που αφορά την ε, αδυναμία έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελα να τονίσω πως οτιδήποτε αφορά πιθανή έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ε, έχει τεθεί, δεν γνωρίζουμε κάποιο τέτοιο αίτημα μέχρι στιγμής, αλλά εάν υπήρχε τέτοιο αίτημα, αυτό βεβαίω θα γινόταν πάντα με τη συνένεση του ε, εν λόγω κράτου μέλου του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ πέρα. Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 28 τη απόφαση, ένα άτομο το οποίο έχει παραδοθεί ε, δυνάμει ενός Ευρωπαϊκού εντάλματος Σύλληψη δεν θα εκδοθεί σε τρίτο σε τρίτο κράτος χωρίς την συνένεση του κράτους μέλους που παρέδωσε το άτομο αυτό. Αυτό για να στονίσω την νομική βάση του θέματος, αλλά βεβαίως το θέμα είναι υποθετικό, γιατί τίποτα συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες, καταρχήν ο κύριος Δίας Δεμέρα, εξ του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μένα το ένταλμα σύλληψης είναι βασικό μέσο για να καταπολεμήσουμε την οργανωμένη εγκληματικότητα και την τομοκρατία, καθώς και άλλες μορφές εγκλήματος. Είναι ένα διαπιστευμένο μέσο και ο ακρογωνιαίος λήθος της συνεργασίας και της πρώτης υλοποίησης του ποινικού δικαίου μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας αναγνώρισης. Βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι κάτι το πολύ χρήσιμο. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε ότι είναι ένα ευάλωτο μέσο. Γιατί όπως είπε και η Επίτροπος Ρέντινγκ, υπάρχει μεγάλη ευαλωτότητα όχι μόνο από την έκθεση της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2011 αλλά και από τις προγενέστερες εκθέσεις ιδιαίτερα του 2006. Βασιζόμαστε σε δύο βασικές αρχές. Το ένταλμα έχει δύο πτυχές, την έκδοση και την παράδοση ημί. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι ένα σκόπιμο μέσον 54.000, από τις οποίες είχαμε 2.000 εκτελέσεις. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε να υπάρχουν μεγαλύτερες δικαιοδοτικές εγγύσεις μεταξύ της έκδοσης και της απόρριψης ή της έκδοσης, της παράδοσης. Έχει βεβαίως μεγάλη σημασία να δούμε και το θέμα της αναλογικότητας. Γι' αυτό με χαρά άκουσα την Επίτροπο Ρέντινγκ να αναφέρει ότι θα προαπαιτηθεί από τα κράτη-μέλη η αρχή της αναλογικότητας και ότι θα πρέπει να, λάβει, να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη και τα πτέσματα, τα μικροεγκλήματα. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε ένταλμα στοιχίζει 25.000 ευρώ στο δημόσιο αυτό ανέφερε ένας Ιρλανδός δικαστής. Και θα ήθελα να πω σε αυτό τον δικαστή ότι δεν το πιστεύω. Θα πρέπει να μου πει ποια είναι τα στοιχεία για να φτάσει σε αυτό τον υψηλό αριθμό. Νομίζω ότι το ένταλμα θα πρέπει να παραμείνει, να ισχύει με βάση τις προπετούμενες εγγύσεις. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μία ε, μπλε κάρτα από τον Earl of Dartmouth. Κύριε Ντεμέρα, δεχόσαστε την μπλε κάρτα. Ο κύριος Ντάκμοθ. Ε, Ο κύριος Διάς γνωρίζει πως η... υπεγράφει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας το 2003 συμφωνία γρήγορη έκδοση πολύ πρώτου ευρωπαϊκού Εντάλματο σύλληψης. Και μήπω θα έλεγε πως αυτό αποτελεί καλύτερο μέσο αντιμετώπισης ε, του σοβαρού εγκλήματο από το Ευρωπαϊκό Εντάλμα Σύλληψη με όλα τα προβλήματα που μόλις ακούσαμε. No. No. Όχι, αγαπητέ συνάδελφε, πιστεύω ότι το ένταλμα σύλληψης είναι ένα καλύτερο μέσο και πιο ευέλικτο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή εγκληματικότητας που προανέφερα. Ήδη το ανέφερε και η Επίτροπος Ρέντινγκ ότι ένα ένταλμα έκδοσης μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο, να διαρκέσει ένα χρόνο. Ενώ σε 40 μέρες θα πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψη σε ευρωπαϊκή βάση. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλύτερο μέσο για να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. και Δημοκράτων. Πρώτη η κατάσταση είναι σαφής. Ακούσαμε το Συμβούλιο να λέει ότι αν εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όπως πρέπει και όχι όπως έχει γίνει μέχρι τώρα σε τριτεύουσα σημασία περιπτώσεις, τότε θα είναι θετικό. Η Κομισιόν από την άλλη μας έκανε μια σοβαρή έκθεση αξιόπιστη που μας λέει ότι αν μπορέσουμε με αναλογικότητα να χειριστούμε ακόμα και τις δευτερεύουσα σημασίας περιπτώσεις θα μπορέσουμε να συλλάβουμε περισσότερους διεθνείς εγκληματίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από τα στοιχεία που έχουμε τα πρόσωπα υπάρχουν αληθινά προβλήματα στη δική μου εκλογική περιφέρεια τα γνωρίζω, ξέρουμε ποιο θα είναι μεταξύ άλλων και το συμβολικό αποτέλεσμα αυτών των μέτρων. Το προφορικό μας λοιπόν ερώτημα στην ομάδα μου σήμερα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή περνάμε από την έκθεση στη δράση και έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι η έλλειψη αναλογικότητας που δεν πρόκειται να λυθεί από μια μέρα στην άλλη. Έγινε λόγος για δικαστική εκπαίδευση, για το ότι υπάρχει κρίση αξιοπιστίας λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού ελάσσων σημασίας περιπτώσεων αλλά θα μπορούσαν και τα κράτη-μέλη να μας βοηθήσουν χρησιμοποιώντας τις προφυλακίσεις αλλά με τρόπο πιο συστηματικό, πιο οργανωμένο όπως πρέπει δηλαδή. Το σοβαρότερο απ' όλα είναι πώς θα δημιουργήσουμε ισότιμες συνθήκες για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της υπεράσπισης ώστε να υπάρχει και ταχεία και ποιοτική διεκπαιρέωση έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που να καταπολεμά το οργανωμένο έγκλημα όπως θα έπρεπε και να μην τύχει κατάχρηση και χρήση μόνο σε ελάσσονο σημασία περιπτώσει. Αυτή είναι η θέση τη ομάδα μου και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη ξέρουμε ότι ζητούν τη δημιουργία, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργηθούν οι ισότιμες συνθήκες εφαρμογής. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Μπέτεμ. Κύριε Μωράη, την δέχεστε. Ορίστε κύριε Μπάτον. Μίλησες Κλώτη για την για την μη ύπαρξη αναλογικότητας. Ξεχάσαμε όμως κάτι το πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ε, το δικαστήριο να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πριν φάση και δεν μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο πρέπει να εκδοθεί ή όχι. Και πολύ ε, πλήττονται από αυτό γιατί σε μία περίπτωση σε περίπτωση ε, κρίσης εφετείου δεν υπήρχαν στοιχεία κατά αυτού του παιδιού. Η, τα στοιχεία ήταν αντιφατικά και δεν ξέραμε κατά πόσο έπρεπε να εκδοθεί ή όχι. Δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν τα υπόψη το δικαστήριο τα στοιχεία πριν με φάση. Η ερώτηση είναι σαφής και ελπίζω να είναι εξίσου σαφής και η απάντηση. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να γνωρίζει το δικαστικό σύστημα ποια είναι τα στοιχεία. Η περίπτωση του Άντρου Σίμιου, όπως είπε ο κύριος Μπάτεν, ήταν διαδικαστικά προβλήματα σε σχέση με την περίοδο κράτησης και μετά από την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, μετά από αυτή την περίοδο ανέκυψαν προβλήματα, κάτι το οποίο προσπαθούμε να επανορθώσουμε με τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίσπεκ, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. και η προγενέστερη συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ζωηρή. Εδώ όμως η συζήτηση είναι πιο συνενετική. Σίγουρα κανένας δεν αμφισβητεί την αποδοτικότητα του εντάλματος σύλληψης, έκδοσης και ούτω καθεξής για να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα. Όμως το ένταλμα όπως χρησιμοποιήθηκε οδήγησε σε καταχρηστικά μέσα όταν μιλούσαμε για μικροαδικήματα Υπάρχει πληθώρα ε, στοιχείων όπως κλέψιμο ποδηλάτων και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο φυλακίζονται και αθώοι και πολλές φορές δεν μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες αυτοί. Γι' αυτό μίλησα για την ε, επιβολή διασφαλίσεων μέσα στα πλαίσια του εντάλματος σύλληψης και σας άκουσα, κύριε Επίτροπε, σήμερα το απόγευμα για να μιλάτε, να μιλάτε για την βελτίωση του συστήματος, να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη και για τους κρατούμενους βεβαίως. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι κάτι το οποίο κατανοούν πολύ καλά οι πολίτες και είναι μια ε, κρίσιμη δοκιμή για να δούμε κατά πόσα η Ευρώπη μπορεί να παγιώσει την, ε, το δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη. Ο κύριος Ζόμπρο έχει το λόγο εξ ονόματος των συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα νέα κρατημέλη χρειάζονται αποτελεσματικά μέσα για να καταπολεμήσουν το έγκλημα, ειδικά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Και άρα μπορούμε να πούμε πως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης απαντά σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει, ειδικά με βάση το ότι ε, ελευθερία διακίνησης δεν έχουν μόνο οι απλοί άνθρωποι, αλλά και οι εγκληματίες, οι οποίοι δεν πάνε για τουρισμό, αλλά πάνε σε άλλη χώρα για να κάνουν εγκλήματα ή για να διαφύγουν από τη δικαιοσύνη. Οπότε είναι θετικό το ότι έχουμε αυτό το μέσο, αλλά πρέπει και να το παρακολουθούμε, γιατί κάθε νέο εργαλείο έχει τα συν και τα πλήν και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το βελτιώσουμε. Θα έπρεπε να περιορίσουμε την εφαρμογή τους για να μην ε, ασχολούμαστε με πτέσματα. Έχετε μπλε κάρτα από την Μπαρόνι Λάντφορτ. Την δέχεστε? Ωραία. Νομίζω πως ε, ο κύριος Γιόμπρο είναι από την Πολωνία και αναρωτιέμαι Συχνά λέμε πως η Πολωνία είναι ένα παράδειγμα των χωρών όπου δεν υπάρχει πράγματι ε, κάποιο κατόφλι για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πώς θα έπρεπε να έχει κάποια διακριτική ευχέρεια ο εισαγγελέα για την έκδοση ε, ευρωπαϊκού εντάλματος και να μην ε, ασχολείται με υποθέσεις όπως το, λεγό, το γνωστό κλεμμένο γουρνόπουλο. Επίσης να πω πόσο εκτιμώ βεβαίως τους περισσότερους Πολωνούς που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο ε, Λονδίνο. Απλά επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός τους έχουμε πολλά εντάλματα σύλληψη από την Πολωνία. Να υπενθυμίσω πως έχετε 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Λέει Παρακαλώ. Πράγματι, ε, γνωρίζουμε το πρόβλημα αυτό που αναφέρατε. Τα πολωνικά δικαστήρια προσπαθούν να είναι αυστηρά, καμιά φορά παρά είναι αυστηρά, και πράγματι δεδομένου του ότι ζουν αυτή τη στιγμή πολλοί Πολωνοί στο Λονδίνο, ε, υπάρχουν ε, πολλά τέτοια εντάλματα. Γι' αυτό Νομίζω πως θα ήταν χρήσιμο η Κομισιόν να ευθύσει κατευθυντήριες γραμμές για να μην χρησιμοποιείται για πτέσματα το έντελμα. Μάλιστα, τώρα θα ακούσουμε την κυρία Σαρτζεντίνη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από το στόμα που το πήρε η κυρία Λάτφορντ. Ήμουν ε, παρούσα στην Πολωνία στη δίκη του κυρίου Κορτισουκούν αναφέρθηκε το όνομά του ενός Ολλανδού ο οποίος εκδόθηκε στην Πολωνία για μια υπόθεση της δεκαετίας του 1990 ε, και σε λίγες ε, ημέρες ε, μέχρι να λάβουν την απόφαση ο Ολλανδός και ο Πολωνός δικαστής εκλάπει το φάρμακο που έπαιρνε αυτός ο άνθρωπος γιατί πάσχει από την καρδιά του. Οπότε βλέπετε πως οι συνθήκες ε, φυλάκισης ε, σε κάποιες χώρες είναι τόσο άθλιες που δεν μπορούμε να αποστείλουμε ανθρώπους εκεί πέρα και θα έπρεπε να είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή που θα εκδώσει να πει ότι εγώ δεν θα στείλω αυτόν τον άνθρωπο σε απάνθρωπες φυλακές και μπορεί να βασιστεί στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Και όταν ακούω το Συμβούλιο να λέει πως ε, οι χώρες ε, θα πρέπει να φροντίσουν τα των φυλακών τους, πράγματι συμφωνώ, αλλά θα πρέπει ε, να μπορέσουμε να πούμε και πως κοιτάξτε αυτό το θέμα είναι πτέσμα τελείως ασήμαντο και δεν θα εκδώσουμε κάποιον άνθρωπο για κάτι τόσο ασήμαντο. Σας ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Στογιάννοφ ε, έχει ένα ερώτημα με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Το δέχεστε, κύριε Στογιάννοφ. Ευχαριστώ. Υποθέτω ότι μιλάτε για την ίδια περίπτωση που προαναφέρθηκε Μιλάτε για την ίδια υπόθεση. Θα ήθελα κι εγώ να υποβάλω την ίδια ερώτηση. Δεν μου δώσατε το λόγο πριν για να αναφερθώ σε αυτή την υπόθεση. Όταν ε, μιλάτε για τέτοιες υποθέσεις να αναφέρσετε στο όνομα των υποδίκων. Θα ήθελα να αναφερθεί το όνομα του υπόδικου, διότι έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά του. Δεν είναι μυστικό, το είπα και πριν το όνομα. Λέγεται Κορ Ντεσούκουν, ο άνθρωπος. Και υπάρχει και η υπόθεση Χόρχνερ, επίσης Ολλανδός, και ο κύριος Ντεσούκουν, όπως ξέρετε, ε, κρατείται σε άθλιε συνθήκε και ζητάει να αλλάξει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ευχαρίστω θα θέλαμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. κύριε Τριανταφυλλίδη, θα αναλεχθούν κύριε Πρόεδρε για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη και την εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη. Μερικά έχουν ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε μια συγκεκριμένη σημαντική πτυχή, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και διαδικαστικών δικαιωμάτων. Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα τόσο ως άνθρωποι αλλά και ως διάδικοι. Όμως αυτά πολύ συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη. Η προφυλάκηση καθώς και οι συνθήκες κράτησης που ανέφερε ο συνάδελφος Ντένις γιονγκ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι γιατί λαμβάνεται ως δεδομένο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τη χάνουν του ίδιου σεβασμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό σαφώ δεν ισχύει γιατί ορισμένα δικαιώματα ερμηνεύονται διαφορετικά ανά κράτο μέλο, όπω για παράδειγμα το δικαίωμα τη σιωπή, ή απλώ επειδή ορισμένε διαδικασίε διαφέρουν, όπω στην περίπτωση τη διάρκεια των περιόδων προφυλάκηση τι σκοπεύετε κυρία επίτροπε να κάνετε γι' αυτό; θα προτείνετε συγκεκριμένα μέτρα όπως την εισαγωγή μιας ειδικής πρόνοιας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που να επιτρέπει στους δικαστές να εξετάζουν το περιεχόμενο των υποθέσεων όπως γίνεται στο ηνωμένο βασίλειο και στην ιρλανδία ή θα παραμείνουν αυτοί απλοί επιβεβαιωτές αποφάσεων άλλου κράτους μέλους; θα προβλέψετε τη δυνατότητα ακρόασης στον ύποπτο ή κατηγορούμενο μέσω της οποίας ένας δικαστή θα αποφασίζει αν πρέπει ή όχι να αποσταλεί ο συγκεκριμένος στη χώρα που τον αναζητεί για να αποφεύγονται καταχρήσεις όπως η έκδοση για πολιτικά φρονήματα. προτίθεστε να προτείνετε τέτοιου είδους αλλαγές στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για τα δικονομικά δικαιώματα ή μέσω μιας τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης the on behalf of the... Ο Δούκας του Ντάρτμουθ. Στον αγγλοαμερικανικό κόσμο, κύριος στόχος του νόμου είναι η προστασία του κόσμου από αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις. Ενώ στην υπηρετική Ευρώπη, ιδιαίτερα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ, ο νόμος δεν έχει τέτοια προτεραιότητα. Περιττό να το αρνηθεί οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε μπορεί να εκδοθεί, παραδείγματος χάρη υπό το βουλγαρικό νόμο, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αντιταχθεί ένας Βρετανός δικαστής σε μια τέτοια έκδοση. Και η Βρετανική κυβέρνηση επίσης έχει δεχθεί αυτό το ένταλμα που είναι περαιτέρω ζημία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσοι αυτό αποκαλούνται κόμμα των δημοσίων ελευθεριών τελικά καταλήγουν πού, στο να τα σταματάνε όλα στο καλέ. Η Βαρονέσα Λάτφορντ, μπλε κάρτα, χωρίς μικαρόφωνο Ο Δούκας του Ντάρτμουθ γνωρίζει ότι οι φιλελεύθεροι μαζί με τους συντηρητικού στην Άνω Βουλή του Βρετανικού Κοινοβουλίου κατάφεραν το 2003 στον νόμο για την έκδοση που κατέληξε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα να δώσουν το δικαίωμα σε ένα δικαστή να αρνηθεί την εφαρμογή αυτού του εντάλματος αν παραβιάζονται τα βασικά δικαιώματα αυτού του ατόμου. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι δεν προστατεύονται τα ατομικά δικαιώματα στη Βρετανία ακόμη και με αυτό το ένταλμα. Να ζητήσετε αν διαμαρτύρεστε από τα δικαστήρια να εφαρμόσουν το άρθρο 23 του νομοσχεδίου εκείνου. Το γνωρίζει λοιπόν ο Δούξ. από την αρχή με μικρόφωνο. Από όσα είπατε, τίποτα δεν ακυρώνει τις επικρίσεις που εκφράζουμε εμείς. Επίσης, κάνετε απολύτως λάθος αν νομίζετε ότι τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνίας για αυτούς τους ανθρώπους ε, τους εμποδίζουν να καταστρέψουν, να καταστραφεί η ζωή τους. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπρόνζ. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα έχουν ε, ελάχιστα κοινά με τις ακροάσεις περί έκδοσης που προϋπήρχαν από το, προϋπήρχαν το 2003. Γιατί εξετάζονται μόνο 10 σημεία και δεν παίζει κανένα ρόλο η έλλειψη στοιχείων στην έκδοση μία ακόμα και εάν το αδίκημα δεν ε, είναι και στις δύο χώρες ε, αξιόπινη πράξη, μπορεί παρόλα αυτά να υπάρχει έκδοση. Επίσης κάποια νεφελώδη εκεί πέρα, αδικήματα σκέψης, ε, τόσο πολύ αγαπητά στην υπηρετική Ευρώπη, πάρα πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο έκδοσης και οδηγούμεθα σε αυτόματη έκδοση σε αυτά τα άθλια μέρη. Οπότε υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος έκδοσης ατόμου για τις ε, πολιτικές ε, του απόψεις. Αν και εδώ πέρα υποψιάζουν πως κάποιες πολιτικές απόψεις είναι πιο ίσες από τις άλλες. Και μιλάτε για τις ε, τρομοκράτες που θα πρέπει να βρεθούν ενώπι, ενώπιον δικαιοσύνη, αλλά οι κακοδικίες τόσων πολλών ανθρώπων δεν είχαν κανένα στοιχείο τρομοκρατίας. Επίσης ε, το χειρότερο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εκδίδονται χωρίς να έχει υπάρξει κατηγορία. Πρέπει να υπάρξει ξανά η απέτηση έκδοσης μόνο όταν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία διάπραξης σοβαρού αδικήματος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας η οποία εκδίδει. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αντωνέσκο έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη είναι ένα πολύ καλό μέσο για να καταπολεμήσουμε τη διασυνοριακή εγκληματικότητα και τρομοκρατία. Αυτό αφορά και την μεταφορά πολιτών οι οποίοι είναι ύποπτοι για μεγαλύτερα εγκλήματα μέσα στα πλαίσια της διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Αυτό το μέσο όμως έχει χρησιμοποιηθεί και για μικροαδικήματα. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το δυσανάλογο, δηλαδή πολλές φορές εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εκεί που ήταν ιδιαίτερα δυσανάλογο διότι πρόκειται για μικροαδικήματα και αυτό δημιουργεί μεγάλο άχθος για το κράτος που εκτελεί. Η δυσανάλογη χρήση για την καταπολέμηση της διασυνοριακής ε, εγκληματικότητας οδηγεί ορισμένα κράτη να προβούν σε έλεγχο της αναλογικότητας και να δουν κατά πόσο πρέπει να εκτελεστεί ένα τέτοιο ένταλμα. Γι' αυτό θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η μη αναλογική εφαρμογή και αμοιβαιότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ίσως βαθμός εκτέλεσης και από το κράτος το οποίο εκδίδει και από το κράτος που εκτελεί. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει και αυτό το ερώτημα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν ίσοι όροι φυλάκισης έτσι ώστε να μην αμφισβητούνται τα δικαιοδοτικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για όλα τα μέτρα που έλαβε για την ενδυνάμωση του ποινικού και της εφαρμογής του από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε την κυρία Αντωνέσκου. Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ. κυρία Ρέντινγκ, στην πραγματικότητα η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα στοιχεία του ε, μέσου αυτού αλλά νομίζω ότι η διασφάλιση αυτών των βασικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να καταστεί δυνατή αυτή η διασφάλιση τη στιγμή που λαμβάνουμε υπόψη τις καταστάσεις, την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές ή την περίοδο κράτησης όπου υπάρχουν διαφορέ στα κράτη-μέλη. Ως προς την αναλογικότητα και τα μικροαδικήματα, θα ήθελα να σας πω, κυρία Ρέντινγκ, ότι όταν μιλάμε για μικροκλεψιές, ποδήλατα, ε, χειρίδια και ό,τι όλα θέλετε, όλα αυτά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι ανάλογα με την έκδοση ενός ε, μίας έκδοσης εντάλματος σύλληψης. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια βάση την κλοπή μιας γραβάτας ή ενός χειριδίου με, το σοβαρό, με ένα σοβαρό έγκλημα. Γιατί το ζήτημα είναι κατά πόσο πρόκειται για ένα μέσο το οποίο είναι αξιόπιστο. Διακόπτει ο Πρόεδρος, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Η κυρία Χαουτάλα, η οποία επίσης έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ούγκρος εκπρόσωπος εδώ μας είπε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με το ίδιο το ένταλμα. Πράγματι, το πρόβλημα σχετίζεται μάλλον με την πολιτική. Ε, καλύτερα να βάλετε ίσως τα ακουστικά σας, ε, γιατί έτσι θα με ακούτε, θα καταλαβαίνετε μάλλον. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα είναι απλώς ένα σημείο κίνησης. Ε, από την αρχή ήδη είχαμε πει ότι θα εφαρμόζονταν ελάχιστα κοινά πρότυπα, αλλά τελικά δεν ελήφθη υπόψη η αλλαγή που επιφέρει η θέση ενισχύ της ε, Λισαβόνας. Τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδιαίτερα στην υπόθεση Γκρέγκ, μας έδειξαν όμως, μας έδειξαν όμως λέγω, ότι σε ορισμένες χώρες οι συνθήκες κράτησης δεν είναι ίδιες από ό,τι σε άλλες. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα όπως ισχύει και στην περίπτωση της Ευρωζώνης. Το ίδιο ισχύει και με το χώρο Σέγγεν. Πολλές φορές η πολιτική ε, δεν είναι τόσο ταπεινή όσο οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αν κάτι δεν έχει αποδειχτεί δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, ε, Σύλληψης ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλά θετικά και η Επίτροπος Ρέντινγκ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας και να μην εφαρμόζονται άκρητα χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσο πραγματικά είναι σοβαρό το αδίκημα. Γι' αυτό θα θέλαμε σίγουρα ένας δολοφόνος να μην μπορεί να περνάει τα σύνορα, αλλά θα πρέπει πράγματι το ένταλμα να έχει και συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν δικαιώματα και για τα θύματα και για τους εναγόμενους έτσι ώστε να έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, δικαίωμα παροχής, μετάφρασης και διερμηνίας και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις, ε, με τις συνθήκες κράτησης θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της κατάστασης, δηλαδή να αξιολογήσουμε έτσι ώστε και οι φυλακές να έχουν όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ο κύριος Στογιάννουφ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Τα επιχειρήματα όσων ασκούν κριτική στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης τα έχω ξανακούσει από τους συναδέλφους από το πατριωτικό κίνημα. Τα επιχειρήματά μας τότε τα είχαμε τα είχαν χαρακτηρίσει ως αντιδραστικά και ότι είμαστε εχθροί της πρόοδου. Σήμερα από την κυρία Υπουργό άκουσα κάτι το φρικτό. Μας είπε πως η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης υπονομεύεται Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πως μία αρχή πρέπει να ακολουθείτε. Καλύτερα να υπάρχουν ε, κυκλοφορούν ελεύθεροι 10 ένοχοι παρά να είναι στη φυλακή ένας αθώος. Οπότε η απάντηση είναι απλή. Πρέπει να τηρούμε τον νόμο και εμείς το Κοινοβούλιο, ο συνομοθέτης, θα πρέπει να φροντίζουμε να ε, υπερέχει ο νόμος. Ευχαριστώ. Κύριε Γιακολίνο. Το Ευρωπαϊκό Ένταμα Σύλληψης είναι πολύ σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση του αργωνωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Αυτό το συμμεριζόμαστε όλοι. καθώς και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Μιλάμε όμως για επιστοποίηση και ενίσχυση των δικαστικών αρχών διασυνοριακά. Mm. Μας ενδιαφέρει το κόστος έκδοσης, ο χρόνος παραμονής ή αναμονής και θα πρέπει να μην θυγεί η αξιοπιστία των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια αυτής της πορείας. Παράλληλα, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το μέσο να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα κράτη-μέλη όπου θα γίνεται μία διάκριση μεταξύ σοβαρών εγκλημάτων και πτεσμάτων. Και θα ήθελα να πω προς την Επίτροπο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν θα λειτουργήσει ίσως θα μπορεί να αξιολογεί τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών ως προς την έκδοση ενταλμάτων. Χρειάζεται μία εποπτική αρχή. Βεβαίως και συνθήκες κράτησης δεν είναι οι ίδιες στα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει την πράσινη βίβλο για τις συνθήκες κράτησης έτσι ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στα κράτη-μέλη. Να γίνεται λοιπόν εύλογη χρήση του εντάλματος, αναλογική χρήση, να υπάρχει μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεργασία των δικαστικών αρχών, διότι μόνο η ομοιογενής εφαρμογή θα οδηγήσει σε ίσες συνθήκες συμμετοχής. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιακολίνο. Κυρία Καστέξ, ευχαριστώ. Βλέπουμε καθαρά ότι η εφαρμογή του εντάλματος θέτει προβλήματα κράτησης με πολύ ανισότιμες συνθήκες από το ένα κράτος στο άλλο. Σε μερικά κράτη ε, δεν υπάρχει καθόλου αυστηρότητα στο σεβασμό των προτύπων της κράτησης και όλο και περισσότεροι σε όλο και περισσότερα λόγω ακριβώς του εντάλματος κρατούνται άνθρωποι σε κράτος άλλο από το δικό τους επομένως πρέπει να γίνονται σεβαστά, σεβαστές οι αρχές που ισχύουν στο κράτος προέλευσης Πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Τον περασμένο Ιανουάριο με τον συνάδελφό μου Σταύρο Λαμπρινίδη είχαμε καταθέσει μια γραπτή δήλωση όπου ζητούσαμε την εναρμόνιση των προτύπων κράτησης στο σύνολο της Ένωσης και την εφαρμογή εθνικών μηχανισμών ελέγχου, ανεξάρτητου ελέγχου. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Επίτροπε κατά τη συγγραφή της πράσινης βίβλου που θα υποβάλλετε να λάβετε υπόψη σας το θέμα αυτό γιατί σε λίγο θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα κοινό υπόβαθρο όλης της νομοθεσίας μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης νομίζω, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αποδείχτηκε ένα χρήσιμο μέσο καταπολέμησης του εγκλήματος πλέον δεν θα εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα εγκληματίες όπως έκαναν μέχρι τώρα. Παρά τις πολλές επιτυχίες που είχαμε όμως, τα τελευταία αυτά 7 χρόνια κατεδείξαν πως το σύστημα δεν είναι τέλειο και δεν χρησιμοποιείται όπως το είχαμε σκεφτεί αρχικά. Κάποια από τα στοιχεία αυτά τα ακούσαμε στην έκθεση ήδη, δηλαδή δεν υπάρχει πάντα παρόν δικηγόρος, δεν είναι πάντα αξιοπρεπής οι συνθήκες κράτησης ε, και ο καιρός επίσης ε, της έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος της αναλογικότητας. Ειδικά αυτό με απασχολεί πάρα πολύ γιατί συχνά έχουμε συστηματική έκδοση για πτέσματα και άρα υποσκάπτεται και η ε, πρόθεση η οποία υπήρχε. Αναφέρθηκε ήδη το παράδειγμα της Πολωνίας που εκδίδει τα περισσότερα εντάλματα και αυτό γιατί οι αρχές δεν έχουν την δυνατότητα να αναστείλουν τις ε, εθνικές διαδικασίες γιατί υπάρχει κάποιος αυτοματισμός. Οπότε θα έπρεπε πριν από την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος να δούμε το βάρος ε, του αδικήματος, ε, μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μία άλλη διαδικασία, ε, λιγότερο ακριβή αν θέλετε, να γίνει και μία ανάλυση κόστους οφέλους. Οπότε συμπέρασμα θα πρέπει να είναι πως θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους κανόνες στην πραγματικότητα και αναρωτιέμαι τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φως. Ο κύριος Παπα-Νικολάου για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων. Ξεκινάω με την κοινή παραδοχή όλων μας, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση. το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην καταπολέμηση του εγκλήματος συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου και στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας και βεβαίως ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της ένωσης κάτι που συζητάμε έντονα το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με το ζήτημα τη σέγγεν εξασφαλίζοντα ότι το άνοιγμα των συνόρων και αυτό πρέπει να το λέμε δεν αποβαίνει ει όφελο εκείνων που επιδιώκουν να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη. Βεβαίω υπάρχουν και φωνέ διαμαρτυρία και συντάσσομαι και εγώ και με αυτά που είπε ο κύριο Βό και με του συναδέλφου, σε ό,τι αφορά την ελλειπή και μη αναλογική εφαρμογή πολλέ φορέ σε εθνικό επίπεδο. κουβεντιάσαμε και για το κόστο και την αναλογικότητα και όλα όσα πρέπει να εφαρμόζουμε και να ενισχύσουμε το ένταλμα σύλληψη. Όμω, υπενθυμίζω και αυτό το αντιμετωπίσαμε και στην ελλάδα πρόσφατα σε σημαντικές υποθέσεις ακόμη και σήμερα υπάρχουν άτομα που διώκονται για σοβαρά εγκλήματα απάτης και διαφθοράς σε κάποιο κράτος μέλος της ένωσης και εξαφανίζονται ή καταφέρνουν να διαφύγουν και να αποφύγουν τη σύλληψη αξιοποιώντα διαφορετικέ δικονομικέ διατάξει και διαφορετικές ρυθμίσει στα διαφορετικά εθνικά δίκαια επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία σε ό,τι αφορά την αξία του ευρωπαϊκού εντάλματο σύλληψη και σε αυτό τοποθετούμε και ε, το λέω ξεκάθαρα σε σχέση και με όσα είπαν άλλοι συνάδελφοι. Κλείνοντα έχετε δίκιο κυρία επίτροπε πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε την Ιντερπόλ, το σύστημα και να ενισχύσουμε την άντληση πληροφοριών από το σύστημα σέγγεν και βεβαίως όσο γίνεται στενότερη εναρμόνιση των κρατών μελών μεταξύ τους για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική εναρμονισμένη σύγχρονη αντάξια των περιστάσεων που απαιτούν οι καιροί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης στόχευε στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν πρέπει να τη χάνει κατάχρησης από εγκληματίες. Οι πρόσφατες όμως εκθέσεις ε, της Κομισιόν, οι δηλώσεις μάλλον της Επιτρόπου Ρέντινγκ, δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν τα ίδια τη σωστή του εφαρμογή, να μην εκδίδεται αυτόματα, ιδιαίτερα για ελάσσονο σημασία εγκλήματα και παραπτώματα. Όταν ένας δικαστής το ζητάει να είναι δικαιολογημένο για να υπάρχει έτσι ως δυνατόν υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας και θα ήθελα η Κομισιόν να παρακολουθεί εκείνη τυχόν ατασταλίες. Ευχαριστούμε. Ήμουν εισηγητή στο σώμα όταν εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψη το 2001-2 και τότε θα θυμούνται οι συνάδελφοι ότι παροτρύναμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ορίσουν περισσότερες ρήτρε διασφάλισης υπέρ των πολιτών και η Επιτροπή μας είπε ότι θα ορίσει μια οδηγία για τα δικαιώματα των ε, υποδίκων, των ε, εναγωμένων. Δυστυχώς η οδηγία αυτή παρέμεινα στο Συμβούλιο επί πολλά χρόνια. Επειδή υπάρχουν πολλές παραλήψεις, γι' αυτό υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία. Το 2002 βεβαίως το Κοινοβούλιο δεν είχε δικαίωμα συναπόφασης. Όμως θεωρούσαμε ότι το ένταλμα εκινεί το προς τη σωστή κατεύθυνση και όπως ολέχθη είναι ένα πολύ αξιόλογο μέσο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Ανέκυψαν όμως προβλήματα από την κακή εφαρμογή από την άκερη χρήση του εντάλματος για μικροαδικήματα και από απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Όλα αυτά μας απασχολούν και θα ήθελα να χαιρετήσω τους, ε, τους συντάκτες όλων ε, όλους τους εισηγητές που ε, τάχθηκαν υπέρ του εντάλματος σύλληψης. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω πως χρειάζεται λίγη κοινή λογική στην συζήτηση. Πιστεύω πως κάποιο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απαραίτητο για να καταπολεμηθεί το έγκλημα και η τρομοκρατία δεδομένης της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων μεταξύ κρατών μελών, με οποίου είναι και εγκληματίες. Επίσης, θεωρώ πως ο αριθμός των λάθων είναι μικρός αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν είναι ανάγκη μαζί με τα χλώρα, μαζί με τα ξερά να κάνουμε και τα χλωρά. Και θα πρέπει να αλλάξει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα για να συμπεριλαμβάνει μόνο σοβαρά εγκλήματα πάντα με το διπλό αξιόπινο και να σεβαστούμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να έχουμε ρήτρες όπως το Habeas Corpus η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων παρέντε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μετανάστες από άλλα κράτη-μέλη της ε, Ένωσης ε, κατά κανόνα για σοβαρά δικήματα και το UKIP, το οποίο κατά κανόνα θα περίμενε κανείς να είναι υπέρ, τώρα προσπαθεί να κάνει ε, δύσκολη αυτή η δικασία για το Βρετανικό κράτος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ομπερμάιρ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι Είχαμε ευρωπαϊκά ε, εντάλματα σύλληψης ε, για το χειρίδιο όπως ακούσατε, για δύο λάστιχα αυτοκινήτου, για τρομοκρατία ουδής λόγος. Και επιπλέον το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, παρεμβαίνει σε πάρα πολύ σημαντική αρχή ε, και λειτουργία του κράτους που είναι η προστασία των υπηκών του και Βεβαίως υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ανεξαρτήτως της αξιόπινης ε, πράξης, ακόμα και αν αυτή δεν είναι αξιόπινη και στα δύο κράτη-μέλη. Για εμένα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης συμβολίζει πλέον το ευρωπαϊκό κράτος εις βάρος των κρατών μελών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Μάιερ. Τέλος η κυρία Αλπάνο. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης αποτελεί το πρώτο μέσο σύμφωνα με το οποίο υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αδικημάτων και αποφάσεων. Έχει μεγάλη σημασία για να καταπολεμήσουμε τη μαφία και το διεθνές έγκλημα. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπου είμαι και η συγγήτρια, μιλάμε για ορισμένες προϋποθέσεις του εντάλματος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να μας αναφέρει κατά πόσο θα ε, μπορέσει με βάση το άρθρο 2 και 3 της απόφασης πλαισίου θα μπορέσει να άρει την διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Τη στιγμή που δεν υπάρχει εκτέλεση ε, θα, πρέπει να μας πει η Επιτροπή ότι κατά να μας πει Επιτροπή τι προβλέπετε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δικαίωμα του συνεταιρίζεστε μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ε, μαφίας. Η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορώ να πω ότι υπάρχει γενική συμφωνία στο σώμα ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης αποτελεί ένα θετικό μέσο και υπηρέτησε πολύ καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ασφάλειας. Τα αρνητικά στοιχεία αφορούν την εφαρμογή του εντάλματος και θα πρέπει να αρθούν φυσικά. Οι προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άρση των αρνητικών στοιχείων αφορούν τη δοκιμή της αναλογικότητας, όπου θα πρέπει να δούμε να εξετάζουμε τη σοβαρότητα των αδικημάτων, το, την ε, σχέση κόστους-οφέλους από την εκτέλεση και τη διάρκεια της κράτησης. Για να γίνει πιο εύκολη αυτή η δοκιμή αναλογικότητας θα υποβάλουμε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της δοκιμής αναλογικότητας. Επίσης χρειάζεται κατάρτιση για τα επόμενα χρόνια. Είναι ύψης τη σημασίας διότι θα πρέπει να καταρτιστούν οι εισαγγελείς δικαστές και συνήγοροι για την εφαρμογή των, του ευρωπαϊκού δικαίου ως προς τους ύποπτους και τους υπόδικους θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες ε, θα ισχύουν και για το ευρωπαϊκό ένταλμα. Συμφωνώ με τους ε, βουλευτές που τόνισαν το θέμα των συνθήκων φυλάκισης στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να τους αναφέρω ότι την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα εγκρίνει την πράσινη βίβλο για τις συνθήκες φυλάκισης. Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνε για τη διαχείριση συνθήκων διαβίωσης στις φυλακές. Η Επιτροπή όμως θα πρέπει να διασφαλίσει την δικαστική συνεργασία έτσι ώστε να τηρούνται τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Γι' αυτό θα αρχίσει μια δημόσια διαβούλευση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για να εξετάσουμε θέματα κράτησης και αμοιβαία εμπιστοσύνης του Ευρωπαϊκού Δικαστικού και Δικαιοδοτικού Συστήματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες φυλάκισης έχουν μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια της αμοιβαία αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και αποτελούν τη βάση συνεργασίας μεταξύ δικαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν οι δικαστές αρνηθούν μερικές φορές πολύ σωστά να εκδώσουν τους υπόπτους εξαιτία των συνθήκων ε, φυλάκισης στη χώρα υποδοχής, τότε έχουν δίκιο. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές υπάρχει κακομεταχείριση των φυλακισμένων. Υπάρχουν ε, πολύ κακές συνθήκες κράτησης. Και όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για τη δικαστική συνεργασία. Επίσης, πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης έχουν σημασία και οι συνθήκες, και οι συνθήκες φυλάκισης και το διάστημα φυλάκισης. Γι' αυτό μας περιμένει πολύ βαρύ έργο και ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να μπορέσω να βασιστώ και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Τέλος, η κυρία Γκιόρη έχει το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Είναι σαφές πως υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία που λέει πως είναι θετικό το ότι έχουμε ένα σύστημα συνεργασίας των δικαστικών αρχών, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Το σύστημα λειτουργεί, δεν είναι τέλειο, πρέπει να βελτιωθεί. Και Πρέπει να σας πω πως βεβαίως είμαστε έτοιμοι για πιο αποτελεσματική χρήση και καλύτερη εφαρμογή. Και βεβαίως συμφωνώ λάθη, συλλήψεις αθώων, όλα αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε και νομίζω πως η καλύτερη εφαρμογή είναι προς το συμφέρον όλων μας. Να γίνω πιο συγκεκριμένη για τα δύο ε, εκρεμή ζητήματα που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα για την αναλογικότητα. Να ξεκαθαρίσω πως ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί να εκδοθεί για δικηματα τα οποία ε, επιφέρουν ε, φυλάξη τουλάχιστον 12 ε, ετών ή για εκτέλεση ε, ε τουλάχιστον 4 μηνών με βάση και την ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1957 για την έκδοση. Νομίζω αυτό αρκεί. Στην πράξη βεβαίως ε, ανακαλύψαμε πως στην περίπτωση λίγων χωρών υπήρχαν ε, παραδείγματα έκδοσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων για ίσονος σημασίας αδικήματα καθώς ήταν πρακτική ε, να εκδίδεται μαζί με το εθνικό και ευρωπαϊκό ένταλμα Οπότε θεωρώ πως θα πρέπει το ακριβό αυτό σύστημα που είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα να χρησιμοποιείται για σοβαρότερα δικήματα. Οπότε ε, αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήταν σωστό τώρα όσον αφορά τις συνθήκες φυλακές. Τα κρατημέλη έχουν μια γενική υποχρέωση να διασφαλίζουν πως ε, οι συνθήκες φυλακές είναι αξιοπρεπείς και δεν αποτελούν απάνθρωπη συμπεριφορά και μεταχείριση όπως αναφέρει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Στην περίπτωση κράτησης ανθρώπου κατά παράβαση των βασικών του ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί αυτός να στραφεί στα εθνικά δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν ξέρω εάν το άρθρο 85 της συνθήκης αποτελεί νομική βάση για ε, να δραστηριοποιηθεί κανείς όσον αφορά το επίπεδο κράτησης στις φυλακές αλλά βέβαια αναμένουμε και τη σχετική πράσινη βίβλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγγέρη. Ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν μέρος στην συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα η οποία τελείωσε.